Όταν σας λέω μιλήσαμε με ειλικρίνεια, ε, πραγματικά σας το λέω γιατί οι Σκοτσέζοι μιλάνε πάντα με ειλικρίνεια. Ο κύριος Λαβία όμως έχει δίκιο ότι πρέπει να προχωρήσει η ψηφοφορία. Ε, γιατί τώρα ξέρουμε ε, περί τίνος πρόκειται και ποιο είναι το διακύβευμα. Έχουμε τον ε, κατάλογο ψηφοφορίας και υπάρχουν αντιπροσωπείες, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι ξέρουν ποιες θα είναι οι key votes και εν πάση περιπτώσει αρκετά κράτησε η προετοιμασία και αυτό το μεγάλο ταξίδι τώρα πρέπει να γίνει η ψηφοφορία. Και επομένως κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε τίποτα άλλο και να προχωρήσει η ψηφοφορία. Thank you very much. Jan. Uh, Πρόεδρος, δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση. Γι' αυτό, Πίτερ, δύο λόγια μόνο αν θέλεις να πεις. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Ντάνκεν για όλα αυτά που έκανε και όλους όσοι βοήθησαν και το βρίσκω πάρα πολύ καλό που ψηφίζουμε γιατί κατ' ουσίαν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ θέλω βέβαια να πω και κάτι άλλο, να ξεκαθαρίσω κάτι για την δική μου την πολιτική ομάδα γιατί υπήρξε μάλλον ε, κάποια παρεξήγηση στον κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, ε, το ΕΛΚ έχει στη σελίδα 7 στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, την πρότασή του και θέλω να πω ότι εμείς είμαστε κατά των τροπολογιών που, έχουν, ε, που ξεκινάνε από το 211 μέχρι το 216. Για μας αυτά είναι key votes και η 217, η τροπολογία 217 ε, από την Κούτελαν και από άλλους 13 ε, ε, βουλευτές των σοσιαλδημοκρατών. Αυτό δεν μας αρέσει. Έχουμε κοιμίων, αλλά δεν είναι key vote. Ως εκ τούτου, εμείς όπως σας είπα θέλουμε να υπερψηφίσουμε. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε κάποια σύγχυση. Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό για μας δεν είναι key vote και ίσως και για κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες αυτό να είναι απόφαση κρίσιμη. Πολύ ωραία. Θέλω να σας πω ότι τα ουγγρικά ε, είναι στο 13. Okay. Do you want to take the floor? θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Να ευχαριστώ όλους ε, και τον κύριο Ντάνκεν και την Λίζα. Το θέμα της ψηφορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ψηφίζουμε. Πρόεδρος, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία πρέπει να σας πω ότι υπήρξε κάποιο λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας και Ήτρε 37, παράγραφος 56. Όχι, λάθος. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ξαναλέω. Ήτρε 37. Καλύπτεται από την συμβαστική πρόταση 13. Δεν θα ψηφίσουμε για την Ήτρε 37 ε, έχει γίνει κάποιο λάθος ε, στον κατάλογο, αλλά τι να κάνουμε, λάθη ανθρώπινα. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι έχετε όλοι μπροστά σας ε, την κάρτα σας. αν έχετε την καλοσύνη να την χρησιμοποιήσετε και όλες, να την βάλετε στην εισδοχή, γιατί σήμερα ε, χωρίς την κάρτα σας τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Κάποιος δεν έχει την κάρτα του. Α, τη βρήκατε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ψηφίζουμε τώρα για τη τροπολογία, τροπολογία 80. Υπέρ παρακαλώ. Κατά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 Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Κι άλλος ένας. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 και 181 ταυτόσημες υπέρ παρακαλώ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 184 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την τροπολογία 19 της εισηγήτριας υπέρ γιατί 19 ψηφίζουμε. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθηση παρακαλώ. Έχουμε δύο από που περισσεύουν. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και άλλη μια ανακοίνωση. Τα σουηδικά είναι στο 20. Δεν είμαι εκφωνητής, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνω. Λοιπόν, ψηφίζουμε για τη 206. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 207 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 208 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για τη 209 υπέρ, κατά, Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Πάμε στην 210, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 211, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ΔΕΒΕ 15 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται, η 215 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 216 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθρηση παρακαλώ για τη 216. Ψηφίσατε όλοι ε, έκλεισε η ψηφοφορία, απορρίπτεται η τροπολογία. Κοιτάξτε, έχει απορριφθεί αυτή η τροπολογία. Δυστυχώς δεν άκουσα με παρατηρήσει είναι εκτός μικροφώνου. Use the mic, please. There's no interpretation when it's off mic. Votiamo il 217. Για τη 217 ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική παλήτηση. Εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ παρακαλώ τη συμβαστική 4, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για τη συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 255 ε, συναδέλφου Ικάουτ. Υπέρ παρακαλώ. Αϊκχάουτ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 17 παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 655 και 656 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Avete Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την συμβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για τη συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Πάλι τώρα αφήνουμε αρκετές τροπολογίες και πάμε στην τροπολογία 23 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε για τη συμβαστική υπεριθμόν 7 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ψηφίζουμε για την τροπολογία 300 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται Φαντάζομαι ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την συμβαστική υπαρτιμόν 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πρέπει να ψηφίσουμε για την 353 και 360 Linen που είναι ταυτόσιμες τροπολογίες. Φαντάζομαι τα έχετε βρει στον κατάλογο ψηφοφορίες που έχετε μπροστά σας. 353 και 360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται και οι δύο. Και ψηφίζουμε 358 για την 358. Μπέλετ, Γκάμπουλς και των υπολείπων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 355. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 345. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 359. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική παλίτευση, εφόσον επιθυμείτε. ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά και τώρα Ψηφίζουμε για τις ε, τροπολογίες 352, 363, 364, 365 που είναι ταυτόσιμες λίγο πολύ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εδώ από την πλευρά μας να δούμε τι έχετε ψηφίσει. Γιατί σήμερα έχουμε κάποιες ομάδες που κάθονται δεξιά και σήμερα, αλλά συνήθως καθόντουσαν αριστερά. Οπότε μας μπέρδεψε. Πάμε στο 366. Υπέρ κατά, άποχες, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Πάμε τώρα στο συμβασμό 10. Συμβασμός 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία, στην τροπολογία 408, Γκούτλαντ και άλλοι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 446. Γκούτλαντ και άλλοι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 447. Πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό 13. υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Συμβασμός 15. Υπέρ του 15 Πρόεδρε. Πάμε πολύ γρήγορα. Πάρουμε, πάμε πολύ γρήγορα. Μπορείτε να επιβραδύνετε πολύ λιγάκι, γιατί δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. Okay. Now we are going to vote. Ας ψηφίσουμε το συμβιβασμό 15. Είναι στην ίδια σελίδα. Στην ίδια σελίδα είναι και οι τρεις. Υπέρ του συμβιβασμού 15, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 460 του Λίζε. Στο δικό μου κείμενο είναι σελίδα 34. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Και τώρα ψηφίζουμε. Στη σελίδα 38, στο δικό μου κείμενο τουλάχιστον, την τροπολογία 508. 508. Γκούτλαντ και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 509. Λίζε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα. Σελίδα 52. Στη σελίδα 52 ψηφίζουμε τις τροπολογίες 60 και 61 του εισηγητή μαζί. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Και τώρα. Ήτρε 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 666 υπέρ. Κατά. Α, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα φοφορίας. Εγκρίνεται. 667 υπέρ. 667 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 668 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 669 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 670 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 671 και ήτρε 34 που είναι πανομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 676 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες 65 και 66 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Votiamo adesso... Ψηφίζουμε. Εξήντα και εξήντα οχτώ. Όχι. Όχι, λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε την 681. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 682-683 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 684 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 685 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69, 70 και 71 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 686 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 687 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 και 73 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ψήφιση της τροπολογίας 688 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για την συμβιβαστική 16. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μήπως ε, δεν πρέπει να ψηφίσουμε 37. Δεν θα ψηφίσουμε για αυτήν. Το είπε. Στην αρχή της ε, ψηφοφορίας και πριν αρχίσει η ψηφοφορία είχα εγγύλει ότι καλύπτεται η Ήτρε 37 από την συμβιβαστική 13. Επομένως δεν θα ψηφιστεί η Ήτρε 37. Αυτή ήταν η τεχνική ανακοίνωση που έκανα στην αρχή. Περνάμε επομένως τώρα στην ψήφιση στις 7.17 μαζί με την ΔΕΒΕ 26. Στην ε, ε, σελίδα 60, σύμφωνα με την δική μου, με το δικό μου κατάλογο ψηφοφορίας, υπέρ, 717, ΔΕΒΕ 26, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 719 και την ΔΕΒΕ 27 από κοινού, υπέρ, κατά, αποχέσε απορρίπτεται. 718 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 720 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 28 μαζί με την 722 και την 723 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 7.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.27, 7.28 από κοινού, διότι είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 83 Κονέτσκνα υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Είμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου. ΔΕΒΕ 4. Ποιος είναι υπέρ της, της τροπολογίας ΔΕΒΕ 4. Κατά. Α, απορρίπτεται. Αποχές, συγγνώμη ξέχασα λίγο πρόεδρος. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 100, μινέρ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 103 και DV11 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 110, ε, Λίζε. Υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με διαφορά μιας ψήφου. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 137 Γκούτελαντ και λοιπή. 137. Στη σελίδα 67 στον κατάλογο ψηφοφορία που έχω εγώ. Λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154, τροπολογία 154 Βυσνιεύσκα Πιέκα. Υπέρ. Κατά. Κα, αποχές απορρίπτεται. Τώρα βρισκόμαστε στην τελευταία σελίδα του καταλόγου ψηφοφορίας που έχω τουλάχιστον εγώ ως πρόεδρος και ψηφίζουμε την τροπολογία 171 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίζουμε τώρα την ε, Ήτρε 15. Ήτρε 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην τροποποιημένη έκθεση, για την τροποποιημένη έκθεση. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα. Πάντα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή, σε όλους τους σκιώδεις για την εργασία την οποία έκανα και δεν έχουμε άλλα σημεία στη μέσα διάταξη. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, μη φεύγετε, μη φεύγετε. Sorry. Miss Dornano to have the floor. Έχετε τον ε, λόγο, κύριε Τζορδάνο Εβάσκες. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μας δεν ε, συμφωνεί με αυτή τη μεταρρύθμιση, την οποία θεωρούμε πολύ επικίνδυνη, πέρα από τις καλές περιβαλλοντικές προθέσεις ή πίσω από τις καλές προθέσεις. Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου είναι πολύ καλή πράξη, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος των ε, βιομηχανικών θέσεων απασχόλησης. Η συντηρουργία, ας πούμε, ήδη ε, υπόκειται σε έναν αμήλικτο ανταγωνισμό από χώρε όπω η Κίνα. Τη στιγμή που έχουν μια σημαντική θέση στον τομέα αυτό, ε, οι χώρες αυτές όμως δεν σέβονται κανέναν περιβαλλοντικό κανόνα. Επιπλέον η ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρος των κυρίαρχων κρατών μελών δεν νομίζω ότι γίνεται σεβαστή σε αυτήν την έκθεση. Επίσης, σφετερίζονται πολλά δικαιώματα ε, διάφορες οργανώσεις όπως παραδείγματο χάρη, ε, συγγνώμη, δεν γίνονται σεβαστές, ε, σεβαστά τα δικαιώματα της α, Διεθνούς Οργάνωσης Αλίας ή Αεροπλοείας κτλ. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ όλων των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να υποκαταστήσουμε αυτές τις οργανώσεις. γι' ακριβώς τους λόγους, καταψηφίζουμε αυτό το κείμενο, αυτές τις τροπολογίες. Είναι μια δήλωση ψήφου αυτή, έτσι. Από ό,τι είχα καταλάβει, για το άρθρο 56.3, εκεί με βάση αυτό το άρθρο ήθελα, θέλατε να ζητήσετε το λόγο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνατε, αλλά τέλος πάντων.